προτάσεις ε, για την ε, διεξαγωγή ψηφοφορίας. Αυτές ήταν ε, οι ανακοινώσεις του Προέδρου. Μπορούμε τώρα να περάσουμε στα σοβαρά θέματα, δηλαδή στην διάταξη των εργασιών που έγινε δεκτή από τη συνδιάσκεψη των Προέδρων στη συνεδρίαση της 5ης 10 Σεπτεμβρίου με βάση το σχετικό άρθρο του κανονισμού και έχετε λάβει αυτή την διάταξη των εργασιών, το τελικό σχέδιο της ημερήσιας διάταξης. Βλέπετε ότι το πρόγραμμα μας ε, είναι πολύ σημαντικό. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τις ακροάσεις ε, των Επιτρόπων και θα ψηφίσουμε σήμερα για τις ε, εγκρίσεις αυτών των διορισμών. Επίσης αύριο θα ακούσουμε την ομιλία για τις ε, πολιτικές και τεχνικές προτάσεις ε, ε, για την επόμενη κοινοβουλευτική, για την επόμενη θητεία του πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επίσης έχουμε τις προτάσεις του, της Σουηδικής Προεδρίας και σήμερα και την Τετάρτη θα μιλήσουμε και για τις αντιπροσωπείες. Το Συμβούλιο θα μας προτείνει και τον κανονισμό για το 2000, τον προϋπολογισμό για το 2010. Βλέπετε ότι η διάταξη των εργασιών μας είναι υπερφορτωμένη, αλλά ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Θα συζητήσουμε λοιπόν όλα τα θέματα με τη σειρά, κύριε Πρόεδρε. Τώρα θα έρθω στο σχέδιο μέρησης διάταξης. Απλώς έκανα κάποιες παρατηρήσεις και για κάθε σημείο μπορώ να σας δίνω το λόγο. Καταρχήν, για το σχέδιο της Δευτέρας, για το σχέδιο μερίσης διάταξης της Δευτέρας, για σήμερα δηλαδή. Υπάρχουν παρατηρήσεις για τις σημερινές εργασίες. Δεν βλέπω παρατηρήσεις, οπότε εγκρίνεται το σχέδιο μερίσης διάταξης της Δευτέρας. Ο κύριος Γκόλνης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, εξαιρετικά λακωνικός θα είμαι. Θέλω να υπενθυμίσω τον κανονισμό ε, σε ό,τι αφορά τη διάσκεψη των Προέδρων. Ε, η διάσκεψη των Προέδρων, όπως είπατε και εσείς, Πρόεδρε, αποφασίζει την ημερήσια διάταξη. Ο κανονισμός λέει ότι η διάσκεψη των Προέδρων, που αποτελείται από εσά και από προέδρους των πολιτικών ομάδων και από έναν εκπρόσωπο των μη εγγεγραμμένων, αποφασίζουν. Αυτή τη στιγμή ο εκπρόσωπο των μη εγγεγραμμένων δεν έχει υποδειχθεί ακόμα. Κάποιοι βουλευτές μη εγγεγραμμένοι σα έγραψαν για αυτό το θέμα και είμαστε στη διάθεσή σας να συναντηθούμε. Θα θέλαμε, κύριε Πρόεδρε, να συγκαλέσετε τη συνεδρίαση όλων των μη εγγεγραμμένων βουλευτών, ούτω ώστε με βάση τον κανονισμό να εκλέξουμε τον εκπρόσωπό μας στη διάσκεψη των Προέδρων. Ούτω ώστε και η διάσκεψη των Προέδρων να παίρνει τις αποφάσεις ε, με απαρτία. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την παρατήρηση και μάλιστα στη διάρκεια αυτής της συνόδου θα έρθω σε επαφή μαζί σας και με τους άλλους συναδέλφους για να διευθετήσουμε αυτό το ζήτημα. Σας ευχαριστώ και παραλαμβάνω εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη της Δευτέρας. Προχωρούμε στην Τρίτη. Σε σχέση με την ημερήσια διάταξη της Τρίτης υπάρχουν παρατηρήσεις. Μόνο για την Τρίτη παρακαλώ. Δεν υπάρχουν παρατηρήσεις για την Τρίτη, οπότε εγκρίνεται και το σχέδιο μερίσης διάταξης Τρίτης. Τετάρτη. Υπάρχουν παρατηρήσεις για την Τετάρτη. Ο πρόεδρος Κομπεντήτ. Αγαπητοί συνάδελφοι, η διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε με ψηφοφορία να βάλει στην ημερήσια διάταξη της Τετάρτης την εκλογή και το διορισμό του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα γίνει μια συζήτηση την Τρίτη το απόγευμα για τις προτάσεις του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εμείς προτείνουμε να αναβάλουμε την ψηφοφορία για την εκλογή του Προέδρου της Κομισιόν για τον απλούστατο λόγο ότι σε 22 μέρες θα γίνει το δημοψήφισμα της Ιρλανδίας. Αυτό το δημοψήφισμα είναι πολύ σημαντικό για την αποδοχή ή την άρνηση της συνθήκης της Λισαβόνας. Σήμερα με βάση μια σφιγμομέτρηση που έγινε, ε, το 62% των Ιρλανδών σκοπεύουν να ψηφίσουν ναι. Νομίζω ότι θα πρέπει να σεβαστούμε την ψήφο των Ιρλανδών. Είτε είμαστε υπέρ ή κατά της Λισαβόνας, δεν έχει σημασία. Το να διορίσουμε ένα πρόεδρο με βάση τη συνθήκη της νίκαιας, ενώ έχουμε τη δυνατότητα, τουλάχιστον όσοι είναι υπέρ της Λισαβόνας, να έχουν μια κομισιόν και έναν πρόεδρο της Επιτροπής που θα διοριστεί με βάση τη συνθήκη της Λισαβόνας μας φαίνεται παράλογο. Για 21 μέρες μόνο και μόνο να κάνουμε νωρίτερα το διορισμό. Τον Οκτώβριο θα ξέρουμε περί τίνος πρόκειται. Ο Πολωνός πρόεδρος δήλωσε επίσημα ότι θα υπογράψει την Λισαβόνα μετά το δημοψήφισμα της ε, Ιρλανδίας. Και το Συνταγματικό Δικαστήριο της Τσεχίας είπε ότι θα αποφασίσει για τις δύο προσφυγές εναντίον της ε, Λισαβόνας, γιατί την τελευταία φορά ομόφωνα είχε πει ε, το Συνταγματικό Δικαστήριο ότι η Λισαβόνα ήταν συνταγματική. Επομένως, ο πρόεδρος της Τσεχίας αυτή τη στιγμή επικυρωθεί η Λισαβόνα από την Πολωνή, από την Τσεχία και την Ιρλανδία να πει όχι. Τελειώνω, Πρόεδρε. Είναι θέμα ταυτότητάς μας για αυτό το ζήτημα. Αν δεν μου δώσετε δύο λεφτά για να σκεφτούμε, νομίζω ότι θα παίξουμε το ρόλο μας ως κοινοβουλευτικοί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σας παρακαλώ. Να μην πούμε ναι ή όχι για τον κύριο Μπαρόζο. Να τον διορίσουμε μετά το δημοψήφισμα των Ιρλανδών. Ας περιμένουμε 21-22 μέρες. Ε, Κύριε Πρόεδρε, δεν ήθελα να διακόψω την ομιλία σας, γιατί όπως ξέρετε τέτοιες ομιλίες ε, υπέρ ε, ενό ψηφίσματο ε, διαρκούν κανονικά ένα λεπτό και η δικιά σα διήρκεσε δυόμιση λεπτά. Βέβαια, ξέρω ότι είναι πολύ σημαντικό το θέμα για σας, αλλά θα ήθελα όλοι οι νέοι ευρωβουλευτές στην αίθουσα να αντιληφθούν ποιοι κανόνες ισχύουν και ότι ισχύουν για όλους. Ακόμη και για τους προέδρους, γιατί όταν υπερασπίζεται κανείς ε, μια πρόταση έχει μόνο ένα λεπτό. Εγώ παρόλα αυτά δεν σας διέκοψα, παρόλο που μακρηγορήσατε, αλλά τέτοιου είδους παρεμβάσει παρακαλώ να περιορίζονται στο ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει ο πρόεδρος Σούλτς. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο συνάδελφος Κον Μπεντίτ ε, έδωσε συνέχεια σε ένα αίτημα που η ομάδα μου στην διάσκεψη των Προέδρων την προηγούμενη εβδομάδα είχε θέσει. Αυτό το αίτημα το θέσαμε επειδή πιστεύουμε ότι λιγότερο είναι το θέμα του δημοψηφίσματος στην Ιρλανδία ή και του συνταγματικού δικαστηρίου της Πράγας αλλά είναι το θέμα της, έλλειψη της έλλειψης της συνεκτικότητας στις απόψεις του Συμβουλίου. Αυτή είναι η βάση αυτής της σύγχυσης στην οποία βρισκόμαστε. Είναι απόλυτα σαφές ότι είμαστε μια κοινότητα νόμου, νομική κοινότητα και πρέπει έτσι να δράσουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση το ενισχύει δίκαιο. Το ενισχύει δίκαιο είναι η συνθήκη της νίκαιας. Δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λοιπόν λύση παρά να εργαστούμε με τη συνθήκη της νίκαιας και για τον Πρόεδρο και όλους τους Επιτρόπους. Αυτό που θέλει το Συμβούλιο είναι ο Πρόεδρος να εκλεγεί, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, με βάση τη συνθήκη της νίκαιας και να γίνει αυτό το οποίο επεσήμανε ο κύριος ε, Κονμπέντιτ πιο πριν. Στη συνέχεια να εφαρμοστεί για τους Επιτρόπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η συνθήκη της Λισαβόνας. Θα έχουμε λοιπόν ένα Πρόεδρο της Επιτροπής που θα έχει εκλεγεί με διαφορετική νομική βάση από την Επίτροπη. Και αυτό εκφράζει ε, παράπονα και ο ίδιο ο πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κάνει λόγο για τι συνθήκε Λισαβόνα που τη χρειαζόμαστε, αλλά που δεν έχει ακόμα αρχίσει να ισχύει. Αυτό είναι η σύγχυση στο Συμβούλιο που υφίσταται και που είναι κάτι το αφόρητο για τον ίδιο τον πρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό θεωρήσαμε εμεί και είπαμε ότι να αναβληθεί η ψηφοφορία μέχρι ότου να συμφωνήσει το Συμβούλιο αυτό που θέλει και να είναι σαφέ αυτό. Γι' αυτό εσεί Πρόεδρε πολύ σωστά Είπατε ότι δύο λεπτά πρέπει να είναι οι παρεμβάσει. Δώστε μου λοιπόν αυτόν τον χρόνο, παρακαλώ. Θεωρούμε λοιπόν ότι η αναβολή για άλλου λόγου από εκείνου που εξήγησε ο κύριο Πεντήτ είναι αναγκαία. Και υποστηρίζουμε γι' αυτόν τον λόγο αυτό το αίτημα. Ευχαριστώ. Ε, ε, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα τώρα να ε, μιλήσει κανείς κατά της πρότασης αυτής. Κατά. Για δύο λεπτά, δύο, το, δυόμιση το πολύ όπως όλοι. Εγώ σέβομαι πάντα το χρονομιλία. Με ξέρετε πολύ καλά, Πρόεδρε. Ούτε δύο λεπτά δεν χρειάζομαι. Καταρχά, δεν καταλαβαίνω τι λέει ο κύριο Κονπεντήτ. Θα έπρεπε κανονικά να ζητήσετε αναβολή τη ε, εκλογή ε, του Προέδρου του Κοινοβουλίου ε, και να περιμένουμε τη Λισαβόνα. Σήμερα ούτω ή άλλω ε, ισχύει το. Εκλέξαμε τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με βάση την νίκαια. Θα ήθελα να εφαρμόσουμε τη συνθήκη τη νίκαια, γιατί αυτήν έχουμε στη διάθεσή μα, μέχρι να τεθεί σε ισχύ η συνθήκη τη Λισαβόνα. βαση τη νικαια θα ζητήσω και κάτι άλλο. Πριν ξαναψηφίσουμε για τον Παρόζο, α σεβαστούμε του κανόνε μέχρι τέλου. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε. Κύριε Κομπεντίτ, να περιμένουμε τη Λισαβόνα και μετά μπορούμε να ψηφίσουμε με βάση τη Λισαβόνα, κύριε Κομπεντίτ. Το βασικό είναι να έχουμε μια επιτροπή, μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό θα ήθελα το Συμβούλιο μετά τις εκλογές της Δευτέρας Οκτωβρίου να διορίσει μια κομισιόν με βάση τη συνθήκη που ισχύει, της Νίκαια. Και την κατάλληλη στιγμή θα συζητήσουμε τη Λισαβόνα. Όταν ο κ. Κομπεντίτ θα πει στον κ. Κλάους να υπογράψει. Όταν ετοιμαστεί ο κύριος Κλάους θα, θα υπογράψει γρήγορα. Και τότε μπορούμε να σεβαστούμε και εμείς στο Κοινοβούλιο τη Λισαβόνα και να ψηφίσουμε και τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τη Λισαβόνα. Γιατί αλλιώς χρειαζόμαστε μια επιτροπή τώρα που να λειτουργεί για την Κοπενχάγη, για τη χρηματοπιστωτική κρίση. Έχουμε ακόμη πολύ χρόνο μέχρι η Κομισιόν και οι Επίτροποι να είναι έτοιμη και να συγκροτηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό θα ήθελα, Πρόεδρε, να ψηφίσουμε την Τετάρτη για τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ωραία, ακούσαμε προτάσεις και υπέρ ε, του πρόταση υπέρ της πρότασης, δύο υπέρ, μία θέση κατά της πρότασης. Αυτοί είναι οι κανόνες να ακούγονται θέσεις και υπέρ και κατά των προτάσεων. Θα ψηφίσουμε τώρα την πρόταση των Πρασίνων Ελεύθερης Ευρωπαϊκής Συμμαχίας. Θα γίνει ηλεκτρονική ψηφοφορία, ονομαστική φυσικά. Παρακαλώ, άρχιτη ψηφοφορία. Czy wszyscy oddali Ψηφίσατε όλοι. Ωραία. Λίγη ψηφοφορία. Ε, 130... Ψήφισαν 397 ευρωβουλευτές, 135 υπέρ, 248 κατά και 14 ε, απήχαν. Οπότε η πρόταση δεν έγινε δεκτή. Το ψήφισμα απορρίπτεται. Ε, υπάρχουν όμως και άλλοι που ζητούν το λόγο. Εγώ ψήφισα, αλλά το... το... και έχω και μάρτυρες ότι ψήφισα, αλλά δεν άναψε το κουτάκι μου, το φωτάκι. Υπέρ ή κατά Μπορείτε να το πείτε. Ψηφίστε υπέρ ή κατά του ψηφίσματος. Υπέρ, υπέρ. Είναι σημαντικό. Θα πρέπει να χαρακτηρίζουμε τις ψήφους. Ήταν υπέρ η ψήφος αλλά δεν αλλάζει τίποτα στο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Το ψήφισμα απορρίφθηκε. Και κάποιος άλλος ζήτησε το λόγο, αν δεν κάνω λάθος. <coughs> Όχι, κανείς. Ωραία. Ο κύριος Σάιερ. Δεν είμαι εγώ κύριε Σάιερ, αλλού κάθεται. Το ίδιο πρόβλημα είχα και εγώ κύριε Πρόεδρε. Δεν λειτουργήσε το μηχάνημα. Εγώ θα ψήφιζα κατά αν το μηχάνημα λειτουργούσε, αλλά δυστυχώς δεν κατάφερα. Καλώς. Άρα ένα-ένα οι δύο τελευταίοι ψήφοι. Ένα υπέρ, Μία, ένα κατά. Άλλες παρατηρήσεις υπάρχουν? Κάποιος άλλος ζήτησε το λόγο στην θέση 607. Ούτε το δικό μου μηχάνημα ε, λειτουργήσε. Ψήφισα κατά όμως. Αυτή είναι η πρόθεσή μου, να ψηφίσω κατά. Καλώς. Ε, όπως και στα ντέρμπι. Έχουμε προπό 2-1, αλλά το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας δεν αλλάζει. Πάντως... Ε, σας καταλαβαίνω απόλυτα. Ο κύριος Στέρντι. Ο κύριος Στέρντι, και εσείς δεν ψηφίσατε. Mr. President. Yeah. I want to record that my... Ούτε το δικό μου μηχάνημα λειτουργούσε. Εγώ ήθελα να ψηφίσω υπέρ του ψηφίσματος. Υπέρ, μάλιστα. E, Θα ήθελα να λάβω μια απόφαση με βάση τις αρμοδιότητές μου. Υπήρξε σαφής απόρριψη του ψηφίσματος, η τριπτική πλειοψηφία το καταψήφισε. Ζήτησαν το λόγο και άλλοι βέβαια, αλλά υποπτεύομαι ότι είναι και το ίδιο θέμα. Παρακαλώ, κάντε μια γραπτή δήλωση και μπορούμε να αλλάξουμε αντίστοιχα το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας γιατί υπάρχει ηλεκτρονική καταγραφή και θα προσθέσουμε και τις δικές σας ψήφους στο αποτέλεσμα. Αλλά με λίγες ψήφους ε, το τελικό αποτέλεσμα, η έκβαση της ψηφοφορίας δεν τροποποιείται γιατί ήταν τόσο συντριπτική η πλειοψηφία του όχι τόσο μεγάλη απόρριψη του ψηφίσματος που με λίγες ψήφους υπέρ ε, δεν πρόκειται να αλλάξει το αποτέλεσμα. Υπάρχουν παρατηρήσεις για το πρόγραμμα εργασιών της Τετάρτης. Όχι, οπότε εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη της Τετάρτης και περνάμε στην ημερήσια διάταξη της Πέμπτης. Για την Πέμπτη υπάρχουν παρατηρήσεις. Όχι, οπότε εγκρίνεται και, το η ημερήσια διάταξη της Πέμπτης και εγκρίναμε το σύνολο των ημερησίων διατάξεων για την Ολομέλεια αυτή. Μπορούμε λοιπόν να περάσουμε το πρόγραμμα της σημερινής ημέρησης διάταξης. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Αντιπρόεδρο Βιτέλη, τον οποίο και καλωσορίζω εγκάρδια. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα σε όλους. Θα πρέπει να ψηφίσουμε την πρόταση απόφασης για τη σύνθεση την αριθμητική των διακοινοβουλευτικών αντιπροσωπιών. Σηκώστε τα χέρια παρακαλώ.